So, was wir schon mal machen können. Αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε για το σχέδιο οδηγίες επιτροπής που τροποποιεί τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς τα πρόσθετα τροφίμων. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, γενικά είναι, δεν έχουμε προβλήματα αυτά. Υπέρ παρακαλώ του ψηφίσματος. Για τη θρομβίνη, το 14 δηλαδή. Υπέρ. Το ψήφισμα για τη θρομβίνη. Η θρομβίνη, υπέρ παρακαλώ. Ας ξαναρχίσω όμως. Δεν έχουμε όμως λύσει το πρόβλημα με τα μηχανήματα. Και για τα ψευδεπίβρα φάρμακα χρειαζόμαστε τις ε, κάρτες μας. Γι' αυτό περνάω στο σημείο 13. Στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των κλικαντικών. Προσθήκη βόγιας και χείριας θρομβίνης. Γιατί είναι μια απλή ψηφοφορία με ναι ή με όχι δηλαδή. Δεν χρειάζονται οι κάρτες. Ο τεχνικός μας είναι εδώ. Ας κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Ηλεκτρονική δοκιμή. Ας ψηφίσουμε το ψήφισμα για τη θρομβίνη με ναι... Α, όχι, με συγχωρείτε, λέει ο κ. Σοβίσεν, υπάρχει μόνο το όχι στο μηχάνημα, δεν επιτρέπει να ψηφίσουμε ναι. So, not working. Άρα μάλλον δεν δουλεύουν τα μηχανήματα. Er- so, we start again. Ξαναρχίζουμε λοιπόν και ψηφίζουμε την, το ψήφισμα για τη θρομβίνη με τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για τη θρομβίνη το 13 ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Και από φαίνεται λειτουργούν τα μηχανήματα. 31 υπέρ, 21 κατά. 31 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές και εγκρίνεται το ψήφισμα. So, dann äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 10. Και πάω προς τα πίσω τώρα στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 10, στα ψευδεπίγραφα φάρμακα, όπου έχουμε μακροσκελή κατάλογο για τις ψηφοφορίες, τον έχετε λάβει ασφαλώς. Ξεκινούμε. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ συμβαστική. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμών 10 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα μερικά φύλλα και να πάμε στη σελίδα 5, ένα φύλλο, στην τροπολογία 157 της Υπέρ της 157 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17 έχει αποσυρθεί. Ήτρε 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετάφραση στα αγγλικά λέει κάποιος εδώ για να ρωτήσω τους ε, συναδέλφους, τους διερμηνείς της αγγλικής καμπίνας αν υπάρχει πρόβλημα. Με τη διερμηνία μας μας ακούτε, το ξέρουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 21 τη Ήτρε. Υπέρ ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159. Περίγιο Ροδρίγε. Υπέρ. Κατά. αποχή, Απορρίπτεται. Τη Σίτρε 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση, ε? Πέρα τη ψηφοφορία. Ναι, ε, εγκρίνεται όπω σα είπα. Με μικρή πλειοψηφία, αλλά εγκρίνεται. Και τώρα προχωρούμε. Στην 19 η ψηφοφορία θα γίνει σε τμήματα. Το πρώτο υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160. Καταπίπτει. Και 161. Στην 20 τώρα. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Δεύτερο. Ε, παρακαλώ. Ε, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα, στην 162, 163, 25 της Ήτρε, είναι ταυτόσιμα σε τρεις αυτές τροπολογίες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 166, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Έγκρινεται. 32 υπέρ, 22 κατά. Στην 27 η ΣΥΤΡΕ που είναι ταυτόσιμη με την 169, υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Οι 170 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτη 176 στο πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν εβδομήντα τρία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Επορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. 175 ηλεκτρονική επαληθεύση. Πέρασε ο 24 υπέρ, 26 κατά. Τέσσερις αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν εβδομήντα τώρα υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, περάσαμε την Ήτρε 28. Γυρνάμε σε αυτή λοιπόν. Υπέρ. Ήτρε 28. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 και 178 που είναι ταυτόσιμες τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 183, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 της Ήτρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 22 κατά, ε, μία αποχή ε, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185-186 ταυτόσιμες, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. 187, η, η 30 της Ήτρε και η 31 της Ήτρε ταυτόσιμες. Μάλλον η 30 και η 187 υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτονται. Και η 31 τώρα της Ήτρε υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 και 32 της Ήτρες το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η 190 και η 32 της Ήτρες στο δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25. υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίσει και ο μικρός. Μπράβο, ωραία. Σωστά ή λάθος. 191 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 194 έχει καταπέσει. Και θα περάσουμε στην 27 στο πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 199. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. σελίδα 12 τώρα. 214 του κυρίου Πρόντι, υπέρ. 214 Πρόντι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 Τη Σίτρε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Καλά το είδα. 28 κατά, 27 υπέρ. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. 11 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 223 και 224 που είναι ταυτόσιμες τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η 225 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 226 καταπίπτει. Στην 228 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. αποχές επαληθεύουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει και πάμε στη 231 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 232-233 Ταυτόσιμες είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 237-238 ταυτόσιμε στη σελίδα 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. η 240, η E340 και η ΙΜΚΟ 12 που είναι ταυτόσιμες τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 241 και 242 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «249» της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρώ στην επόμενη σελίδα. 248. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 258-259, ΙΜΚΟ 13 και οι τρεις ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 260-261 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Διακόσια εξήντα τρία. Και 264 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 265-266 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 267-268. Όχι, θέλετε να επαληθεύσουμε. Τη 265-266 παρακαλώ. έχει δύο παραπανήσιες ψήφους στο ΕΛΚ τώρα. Συγγνωηθείτε ποιος θα αποσυρθεί. Άλλος ένας. Να, εντάξει τώρα. Πέρασε τις ψηφοφορίες. 30 υπέρ. 25 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρινέται. 268-268. Αυτό σημαίνει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ε, πιο κάτω στη σελίδα 275 του κυρίου Λίσε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...279 πρώτο τμήμα και 280 πρώτο τμήμα ταυτόσιμες και μαζί έχουμε και την έμικο 17 πρώτο τμήμα. Να ψηφίσουμε λοιπόν αυτές. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνονται. ...279 τώρα δεύτερο τμήμα... ...τη 280 δεύτερο τμήμα... ...και τη 278 δεύτερο τμήμα... ...και την ΙΜΚΟ... ...τη 17 της ΙΜΚΟ δεύτερο τμήμα... Υπέρ αυτών των τεσσάρων τροπολογιών παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνονται. 279 τρίτο τμήμα, 283, τρίτο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στη 17 της ΣΥΜΚΟ το τρίτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές. Απόρριπτε 278 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στην σελίδα 19 κατευθείαν. 288 των κυρίων Τρεμόπουλου και Ριβάση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 και 18 τη Ήτρε τώρα, ταυτόσιμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 46 τη Ήτρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση θέλετε. 46 τη Ήτρα. Επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 292 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 της ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 293 και 294 μας υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά στο το επαληθεύσουμε αν θέλετε. Πέρα στις προφορές. Έχουμε μία περίσσια ψήφο από το ΕΛΚ πάλι, παρακαλώ, να αποσύρετε μία κάρτα. Τώρα εντάξει. Απορρίπτεται. 25 υπέρ, 31 κατά. 295 υπέρ. 295. Περέιο Ροδρίγε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 299. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 300. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 301. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 48 της Ήτρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 της Ήτρα και 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 305 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 306-307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 και 309 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά αποχές δεκτή ταυτόσιμες 3.13 ε, και 3.50 υπέρ κατά αποχές δεκτές 3.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.16 και 54 της υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3.17 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3.17 μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. κάτω-κάτω. 3.23 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.23 μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 326, 327 και η 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε στη σελίδα 23 κάτω κάτω Η 360 υπέρ. Κατά. Στην σελίδα 23 τελευταία τροπολογία. Η γραμματεία μου λέει πως όλες οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Γιατί ε, έγινε δεκτή η 19 της ΙΜΚΟ. Οπότε είμαστε στην σελίδα 23 την 60 της ΙΤΡΕ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές δεκτή. 338 τρία, οχτώ μετά, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 3.42 υπέρ κατά δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν είμαστε στην 3.42 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 342 και την Ήτρε 61 μαζί πανεύθες. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. Όχι, είναι σαφές. 31 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Μετά έχουμε την συμβαστική νούμερο 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τρία σαράντα εφτά Κέρμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3.48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 350 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές δεκτή μκο 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 352 και η 367 υπέρ κατά αποχές δεκτή 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 354 και η 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 355 υπέρ κατά αποχές δεκτή 356 υπέρ κατά αποχές δεκτή ή 369 υπέρ κατά αποχές δεκτή 357 ή 370 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 και η 371 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 23 χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΤΡΕ 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 361 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 έχει αποσυρθεί 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμκο 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 75 υπέρ Ήτρε 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή να, να ελέγξουμε Ήτρε 75 Abstimmung beendet. Πέρας της ε, ψηφοφορίας, όχι είναι σαφές. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην 51 και ίδρα υπέρ. Ποιος είναι υπέρ και ίδρα ένα με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Αποχές. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει επόμενη 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ και η 7 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σελίδα 32. Στην 83 της κυρίας Παρβάνοβα είμαστε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Πού, πού είναι αυτό που λέτε. Στην 32 είμαστε. Πρώτα ψηφίσαμε την 83. Εγώ δεν βλέπω καμία 61. Äh, Κύριε Ζέμπερ, καλύπτεται από την ε, συμβαστική 4, οπότε συνεχίζουμε. Του ήμασταν... Ήμασταν στην 85. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86-87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. στην επόμενη σελίδα 84 Μπαρτολότσι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 αποσύρεται Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 και ήτρε 13 υπέρ κατά αποχές δεκτές 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 και ήτρε 15 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε πρώτο μέρος υπέρ ε, πρώτο μέρος με συγχωρείτε επαλήθευση στο πρώτο μέρος, στο πρώτο μέρος. Το επαληθεύουμε. So, alle abgestimmt. Ψήφισαν όλοι. Τριάντα υπέρ ή 21 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ή 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά 101 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε. 101. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα είναι εντάξει. 31 υπέρ 19 κατά ε, σαφές 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 και ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές δεκτές 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 και 122 ταυτόσιμες χωριστή ψηφοφορία από το μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος. Πέρας. 26 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. Καλά κάναμε και έλεγξαμε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οπότε φτάσαμε ήδη στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση της Ματίας Άρχεται η ψηφοφορία. Το, από το είναι ένας παραπάνω. Τώρα είναι εντάξει. Πέρας. Οπότε 51 υπέρ 3 αποχής Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια και ερχόμαστε στην δεύτερη τελική σοφορία, άρχιτη σοφορία. για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 46 υπέρ κατά δύο αποχές. Εξίσου. Σαφές συγχαρητήρια στην Μαρίζα Ματίας για την έκθεση. Συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη. Με τη φαρμακοεπαγρύπνηση τις εκθέσεις της Λίντα Μακάουν. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, είμαστε όλοι σε φόρμα για να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά ψηφοφοριών. Έχουμε δύο εκθέσεις για τη φαρμακοεπαγρύπνηση της Λίντα Μακάβεν. Μία είναι η οδηγία, μία είναι η άλλη είναι ο κανονισμός. Θα αρχίσουμε με τον κανονισμό. Αντίθετα με αυτό προβλέπει λοιπόν η ημερήσια διάταξη, ψηφίζουμε πρώτα τον κανονισμό. Μην μπερδευτείτε, regulation. Έχετε τον κατάλογό σας για τις ψηφοφορίες και αρχίζουμε με την υπαριθμόν 1 τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Βλέπω ότι δεν ε, συμπράττουν όλοι με τον ίδιο, στον ίδιο βαθμό. Είμαστε στον κανονισμό, όχι στο ψήφισμα. Στην τροπολογία 34, για να μην έχουμε μπερδέματα, υπέρ παρακαλώ. 34 κατά τις 34. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Φαίνεται ότι είναι πολλοί εκείνοι που δεν έχουν φέρει τις κάρτες τους, δεν τις έχουν βάλει στο μηχάνημα. Πέρασε τις ψηφοφορίες λοιπόν. Απορρίπτεται 22 υπέρ 26 κατά. Επτά υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 τώρα, υπέρ, υπέρ της συμβαστικής 3. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται συγγνώμη κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 της ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 τη ΣΥΜΚΟ κάτω κάτω στη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 13 τη ΣΥΤΡΕ υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την 13 η σύντροφη, παρακαλώ. Απερίφθη, είναι σαφέ το αποτέλεσμα, εγώ έκανα λάθο. Δεν πρόσεχα. Απορρίπτεται λοιπόν. 48 υπέρ. 48 κατά αποχές. Δεν δουλεύει το μηχάνημα. Μια προφορική τροπολογία μόνο, Πρόεδρε, για τον εντοπισμό ή την αναγνώριση. κομμάτι της ψηφοφορίας ήταν αυτό. Έχει γίνει δεκτό. Στην 47 τώρα ριβάζει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και υπάρχει μια κάπως παράδοξη τυματική ψηφοφορία.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 η γραμματεία μου λέει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε και το δεύτερο τμήμα της ε, πέμπτης τροπολογίας ΣΥΜΚΟ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. μόνο 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. στην επόμενη σελίδα. 61ο τμήμα Μακίνας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 57-58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 τμήμα υπέρ κατά αποχές 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 16 της Σίτρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 ριβαζή και 17 της Ήτρε ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 11 πρώτο τμήμα και τροπολογία 9 πρώτο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. 11 της 20 δεύτερο τμήμα και 9 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. 63 ΕΜΚΟ 12 ή 18 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Μία περίσσια ψήφος από το ΕΛΚ. Απορρίπτεται λοιπόν 25 υπέρ 28 κατά. Κάτω-κάτω τώρα πάμε στην 64. Στην ίδια σελίδα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 και 19 τσίτρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ενοποιημένη τροπολογία 2β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλά, ας επαληθεύσουμε. Ενοποιημένη τροπολογία 2β. Πέρασε σου 20 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Θέλετε παλήθευση στην 70. Άρχεται η ψηφορία. Πέρα στις 30 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Τι ήταν αυτό. Πρέπει να σας πω ότι με την αντιλιά που έχει από τα παράθυρα δεν βλέπω πάντα καθαρά τα χέρια. Ίσως αυτό φταίει. Ε, στην 71 τώρα υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 12 και 73 και 21 της Ήτρε. Ταυτόσιμες είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται, αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Και προχωρούμε στην 72 υπέρ. Κατά άποχες. Εγκρίνεται. 21 της Στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 12 στο δεύτερο τμήμα, 72 στο δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτει άλλη. 74-75 ταυτόσιμες. Υπέρ κατά. Από ποιες εγκρίνονται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παρήθευση. Καλώς. Abstimmung beendet. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Εβδομήντα εφτά. Τώρα. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 78 και 22 της Σίτριπερ κατά αποχές εγκρίνεται 13 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απρέπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μετά πάμε στη λύση Ούλμερ, 82 δηλαδή υπέρ κατά. Αποχές. Απορρέπτεται. 17 της ΣΥΜΚΟ και 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο αλφα Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16-17 ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η πρώτη της ήτρε ήταν μέσα. Στην 20 και δεύτερη της ήτρε τώρα. Υπέρ κατά αποχές ας κάνω μια επαλήθευση Πέρα τις εγκρίνεται ή δύο παρακαλώ τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Στην τέσσερα τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρώ στη συμβαστική υπαριθμών 1. Υπαριθμών 1 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 και 6 της ΣΥΤΡΑ μας υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβασ... Ε, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Στο σύνολο τώρα το σχέδιο της έκθεσης άρχεται η μία περισσία ψήφο στο ΕΛΚΑ. Ξεκολουθείτε τώρα. Τώρα εντάξει. 52 υπέρ, χωρίς καμία ψήφο κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και να δούμε και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με τα ίδια αποτελέσματα. 52 υπέρ, χωρίς ψήφους κατά και αποχές. Συγχαρητήρια, Λέντα. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη Συνεχίζουμε όμως. Μετά τον κανονισμό πάμε στην οδηγία για την φαρ... Κυρία Γιούσο. Πριν ξεκινήσουμε και για να μην διακόψω αργότερα, θα ήθελα να πω ότι αποσύρω την τροπολογία μου 84. Ευχαριστώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 72 και 10 της ΣΥΤΡΕ που είναι ταυτώσουμε Κατά αποχές απορρίπτονται. 75 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτονται. απορρίπτεται. 74-76 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 79 τώρα. Κατά. Αποχές. το. Την 84, η 84 έχει αποσυρθεί. 11 της ήτρε παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 και 82 και η 83 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ, 85 συγγνώμη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 12 της Ήτρα και 88 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτονται 89 ε, και 90 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 13 της Ήτρα παρακαλώ ναι, θέλετε να το 9 και 90 εντάξει Πέρας τις προφορίας. Δεκατρία της ήτρε παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψτε. Ερεντέ, 92, 93, μας υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 95 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ήτρε 14 και 94 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 94 δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 και 95, ή 13-14 δεύτερο τμήμα, δηλαδή και 95 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 94 τρίτο τμήμα, 95 τρίτο τμήμα, 14 τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 95 τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Οχτώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 ψηφίζουν, αλλά 53 ε, είναι οι κάρτε μόνο. Γι' αυτό μερικέ φορέ με την ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν τι κάρτε του. Γι' αυτό βλέπουμε και την απόκληση όταν κάνουμε την επαλήθευση. Εν πάση προχωρούμε. 97 και 14 τη παρακαλώ υπέρ κατά αποχές. 15 Απορρίπτονται. 96 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98, 96 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 τη δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 τρίτο τμήμα, 99 έτσι 15 ταυτόσουμε στο τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 100 παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ καλά. Να ελέγξουμε λοιπόν, να επαληθεύσουμε την 100. Πέρα στις ψηφοφορίες. Το ίδιο. Ενώ έχουμε 56 παρόντες, ψηφίζουν 51. Πέντε είναι αυτοί που δεν έχουν κάρτα τώρα. Απορρίπτεται, βάση περιπτώσει. Κάναμε την Ήτρε και την 95. Ε, γυρνάμε σελίδα λοιπόν. 101-102. Δεν γυρνάμε σελίδα. Στην 3 είμαστε ακόμα. 101-102 είναι ταυτόσιμες. Παρακαλώ υπέρ. υπέρ. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ενοποιημένη τροπολογία του 2α, ε, υπέρ παρακαλώ, κατά εποχές εγκρίνεται. Και έτσι προχωρούμε για να πάμε στη σελίδα 6. 118 ροτ parent, υπέρ. Κατά χέρι εγκρίνεται. Εννέα της ΕΜΚΟ. Και 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120-121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 18 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 122 παρακαλώ. Πέρας. 32 υπέρ, 21 κατά. Υπαριθμών 5 συμβαστική παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσεχή σελίδα 134 μαστάλκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 τη ΣΥΜΚΟ. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 12 της ΙΜΚΟ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 12 της ΕΜΚΟ πρώτο τμήμα. Μάλιστα, να ελέγξουμε. Ποιος το ζητάει. Ελέγχουμε. Την 12η ΣΥΡΜΚΟ πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 25 υπέρ 28 κατά. Πάντω επαναλαμβάνω, αυτά που βλέπω εγώ με τη στρανάταση δεν ε, συνάδουν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πάμε παρακάτω όμω 135, Αγίου Παρανόβα, υπέρ, Περβάνοβα, παρασύνομαι, υπέρ, κατά, Αποχε. εγκρίνεται. 12 δεύτερο τμήμα, 12 τη υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. 12 τη ΣΥΜΚΟ, δεύτερο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 136 και ήτρε 20 μαζί υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 και 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Και η 321 βέβαια ήταν αυτό Η 122 ε, της ε, Ριβάζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 Ριβάζη πάλι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 144. Πέρας. 21 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. 14 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα 25 της ήτρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα στην ενοποιημένη 2β Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι, κερδίζουμε αρκετό χρόνο και προχωρούμε στην ε, σελίδα 11 και στην 16 της ΣΥΜΚΟ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήταν ταυτόσιμη μάλιστα. Όχι, τώρα προχωρούμε και στη 12. Έχουμε ψηφίσει 164, 165 κτλ και οι 17 που είναι ταυτόσιμοι και 166 τώρα. Εδώ είμαστε. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. 167. Πέρας της 6 υπέρ 25 κατά. Εγκρίνεται. Κατόν 68 η Ροδρίγης υπέρ. Κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 168. Πέρασε φοφορίες. Απόλυπτεται. Από τη μία πτέρυγα πέντε συνάδελφοι δεν έχουν μαζί τις κάρτες τους. Τι να πω. Δεκατρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρασε τις προφορίες. Εγκρίνεται. Όχι, όχι, συγγνώμη. 26 κατά. Μάλλον πρέπει να αναλάβει η κόρη τώρα. Έχω κουραστεί. Λίσε Ούλμαρ, 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 14. Η στην 29 πρώτο τμήμα. Κατά αποχές απορρίπτωται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190 καταπίπτει. Και πάμε στην επόμενη σελίδα. 195, 196 και 30 της σύντρα. ταυτόσιμες είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, δεν, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη πια έτσι, ε. 197 Πέρασε προφορίες. <laughs> ναι. Ε, λοιπόν, εγκρίνεται. 27 υπέρ, 24 κατά. 200 της κυρίας Λεπάζ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 της κυρίας Λεπάζ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε πέρας της πληροφορίας. 24 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα φαντάζομαι, αλλά σε παληθεύσουμε. Πέρασε 30 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 17, ημικο 25. Και 219. μας είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 πρώτο τμήμα. 223 πρώτο τμήμα. Αυτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 221 πρώτο τμήμα. Θέλετε να επαληθεύσουμε. 220 πρώτο τμήμα 223 πρώτο τμήμα. Ένας που περισσεύει από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει. 24 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 221, πρώτο τμήμα. 33 της ΙΤΡ, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. «222 δεύτερο τμήμα, ήτρα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται». «224 πρώτο τμήμα, 33 της τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 221 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 223 δεύτερο τμήμα, 220 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε παρακαλώ. 223 και 220. Στο δεύτερο τμήμα και τα δύο. Πέρες φορές. 30 υπέρ 23 κατά. Εγκρίνεται. 225 και 26 της ΣΥΜΚΟ. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 224 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 221 τέταρτο τμήμα και 33 της τέταρτο τμήμα και 224 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 27 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 221 πέμπτο τμήμα, ήτρε 33 πέμπτο τμήμα, 228 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 16 της ηγετρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 221 έβδομο μέρος, 228 δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 33 έκτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 27 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.26 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε μια επαλήθευση του 226 Πέρας. 28 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται 227 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 8 μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 ένατο μέρος 229 ή 33 έβδομο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 29 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. 232 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Ταυτόσημη 239 πρώτο μέρος και 241 πρώτο μέρος υπέρ. κατά αποχές απορρίπτονται και η, η 34 ήταν εκεί μέσα επόμενη σελίδα 241 μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ταυτόσιμες αρκετές Μπουόζι, Ριβάζι, Ντελβό και Ήτρε ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ταυτόσημες ΙΜΚΟ και ΖΟΥΒΕΝ υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ήμκο και ΖΥΒΕΝ. Να επαληθεύσουμε. 29 δεύτερο μέρος και 233 αρχεται η ψηφοφορία. Ήμκο 29 δεύτερο τμήμα και Ζουβέν 233. Πέρας. Κλέρ. Κλέρ, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, αρκετά πιστικό. 234, 235 και 17 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτές. 243 τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 241 τρίτο μέρος ή 334 τρίτο μέρος υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Ήμκο 30 και 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 240 τέταρτο μέρος και 241 τέταρτο μέρος ή 334 τέταρτο μέρος, 239 τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ήτρε 34 πέμπτο μέρο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 236 πέρ. Κατά. άποχε απορρίπτεται. 238 υπέρ. Όχι. Identisch, ja, να είναι ταυτόσιμη. Άρα πάμε στην επόμενη 2.39 τέταρτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 55 υπέρ. 35 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 δεύτερο μέρος β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 τέταρτο μέρος υπέρ κατά εποχές. απορρίπτεται 242 πέμπτο μέρος πέρ. κατά εποχές. απορρίπτεται 242 έκτο μέρος πέρ. κατά εποχές. απορρίπτεται 245 υπέρ κατά εποχές. απορρίπτεται 247 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 31 και 243 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 32 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την ΙΜΚΟ 32. Πέρας. Τσίμα τσίμα ήταν. 26 υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 33 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 249 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή να επαληθεύσουμε την 250. Πέρας. 26 υπέρ, 24 κατά, 2 αποχές δεκτή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 249 δεύτερο μέρος υπέρ. κατά άποχες δεκτή 249 τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 251 υπέρ κατά Ε, τελικά το ΕΛΚ είναι κατά ή υπέρ. Ας επαληθεύσουμε, γιατί βλέπω μόνο τους μισούς. Την 251 λοιπόν. Και πέρασε. 26 με 26 απορρίπτεται και πάλι. 51, όχι 21, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά να ελέγξουμε γιατί είναι 22 πέρας απορρίπτεται 27 έναντι 26 ή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 252 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτρε 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήμκο 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 253 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 δεύτερο μέρος του συγγητή υπέρ της συγγητρίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 35 και 253 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 255 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτεί, 2.56 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 256 πέρασε 27 υπέρ 26 κατά δεκτή. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή 2.58 και ήτρε 38 ταυτόσημες υπέρ κατά να επαληθεύσουμε. ...2.58 και ήτρε 38 πρώτο μέρος. Ψηφίζουμε. ξανά. Α, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ 28 κατά. Απορρίπτονται. 259 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. 27 υπέρ, 26 κατά. Δεκτή. 260 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Abstimmung beendet. Πέρασε. 26 με 26 Απορρίπτεται όμως. Ή 338 δεύτερο μέρος και συνυπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 25 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 25 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται. Ταυτόσιμες 2 68 και η 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 263 Σνέλχαρτ υπέρ κατά αποχές δυστυχώς απορρίπτονται κύριε συνάδελφε ενοποιημένη 4β ποιος είναι υπέρ της 4β κατά αποχές απορρίπτεται 264 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Να επαληθεύσουμε. Την 264. So, 32 υπέρ, 18 κατά. Δεκτή. 265 υπέρ. Α, καταπίπτει. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά ταυτόσημες ΣΥΜΚΟ 36, 267, 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ταυτόσημες 269 ή 339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 266 άντε repair Κατά. Να επαληθεύσουμε. Την 266. Πέρας. 26 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 37 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την Ήμκο 37. Πέρας. 29 υπέρ 24 κατά δεκτή. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. πέρας 31 υπέρ 22 κατά δεκτή περνάμε στα εκτιμώντας 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Πέρας είναι υπέρ 24 κατά δεκτή ή τρένα υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. 29 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Πέρασε. 27 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται. 28 κατά καταπίπτει και ερχόμαστε συμβαστική 4α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 32 πέρας 21 υπέρ 32 κατά απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 2 να επαληθεύσουμε την 35 πέρας 27 υπέρ 27 κατά Απορρίπτεται. Η δύο υπερ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2C υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Επόμενη σελίδα. Συμβαστική 1β υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. Και πάμε στην 51 υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. Οπότε συνεχίζουμε με την ΙΜΚΟ 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 55 και 56 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 6 ήταν μέσα εκεί 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 59 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή κατόπιν περνάμε στην 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 δεύτερο μέρο υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 ή 7 ταυτόσιμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά εποχές να επαληθεύσουμε είναι 65 πέρας 28 υπέρ 26 κατά δεκτή 66 και ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 67 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 67 πέρας 29 υπέρ 23 κατά δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 και ήτρε 9 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε πέρας 26 υπέρ 28 κατά Α, απορρίπτεται Ήμκο 7 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε πέρας. 26 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Νούμερο 7 κατόπιν. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Οπότε ήσασταν φανταστική. Ωραία. Τα καταφέραμε. Περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για ολόκληρη την έκθεση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 49 υπέρ, κανείς κατά μία αποχή και περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης 49 υπέρ 5 αποχές. Συγχαρητήρια στην Λίντα Μακάβαν. Για αυτά τα οποία έκανε για την ασφάλεια των φαρμάκων. Καλά. Τα πήγαμε, οπότε τα ξαναλέμε το απόγευμα στις 3. Α, δεν έχουμε τελειώσει. έχουμε την έκθεση της αντιπροσωπείας ε, για την υπηρεσία χημικών στο Ελσίνκι, την ΕΚΑ, μια σημαντική υπηρεσία για εμάς. So, die Kontaktperson zur ist η Σάτου Χάση είναι η υπεύθυνη για την υπηρεσία αυτή. Äh, θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Σατουχάση να μας πει τα της επίσκεψης στο Ελσίνκι. This came as ε, Είμαι προεκπλήξεως. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν με είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να σας κάνω τον απολογισμό, επομένως δεν είμαι προετοιμασμένη. Θα πω κάποια πράγματα βέβαια. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων εφαρμόζει νομοθεσία η οποία προσπαθεί να αλλάξει πολύ την πρώτερη κατάσταση και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ακούσαμε πολλά πράγματα για τον προϋπολογισμό, ε, οργανωτικά θέματα, θέματα πληροφορικής, IT. Στη συζήτηση μετά την ε, έκθεση ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο έχει θέσει η Επιτροπή μας ε, επανειλημμένος. Και αυτό είναι το θέμα των υποψηφίων ουσιών, του καταλόγου υποψηφίων ουσιών, τα οποία είναι στη διαδικασία της έγκρισης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν περίπου 500 ουσίες οι οποίες δεν είναι ενδιάμεσες της πετροχημικής βιομηχανίας και οι οποίες είναι γνωστό ότι πληρούν ε, τα κριτήρια για, ε, και θεωρούνται ουσίες ε, πολύ επικίνδυνες, CMR, BPT, BBB. Αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των υποψηφίων ουσιών έχουμε μόνο 30 χημικές ουσίες. Η πρόοδος λοιπόν είναι πάρα πολύ αργή και για τους πολίτες ένα σημείο το οποίο είναι σημαντικό και δεν υλοποιείται ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος είναι το δικαίωμα του καταναλωτή να είναι καλά πληροφορημένος στην οδηγία υπήρχε το δικαίωμα του καταναλωτή να ενημερώνεται για τις επιζήμιες ουσίες, αλλά προς το παρόν ε, ε, περιορίζεται η ενημέρωσή του μόνο στις ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο των υποψηφίων προς έγκριση. Οι Επίτροποι ε, Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος, Ποτότσιν και Ταγιάννη, κατέληξαν στο συμπέρασμα και συμφώνησαν επ' αυτού ότι θα πρέπει να γίνει κάποια περαιτέρω πρόοδος και συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο μόνο το 25% των γνωστών ουσιών που έπρεπε να βρίσκονται στον κατάλογο αυτό ε, έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν. αυτό το οποίο διαπίστωσε η αντιπροσωπεία μας είναι ότι το σκεπτικό της Επιτροπής είναι ότι ε, θεωρούν ότι υπάρχουν δύο στάδια στην ομοθεσία. Το να συμπεριλαμβάνονται οι ουσίες αυτές ε, στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών και υπάρχει και ένα επόμενο βήμα που είναι οι αποφάσεις για ουσίες οι οποίες θα περάσουν ε, στην ε, διαδικασία έγκρισης. Θέλουν να γνωρίζουν δηλαδή ότι κάθε ουσία που βρίσκεται σε αυτόν τον κατάλογο υποψηφίων θα φτάσει μέχρι την ε, τελική έγκριση. Ίσως αυτό να είναι κατανοητό από πλευράς υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της νομοθεσίας, όπως σας είπα, είναι το δικαίωμα του καταναλωτή να είναι ενημερωμένος και αυτό κάπου χάνεται στη διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι επίση σημαντικό για την Επιτροπή μας είναι ότι συνειδητοποίησαμε στη διάρκεια της επίσκεψής μας ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων στον οποίο εγώ έχω πάντα πάει ως ε, άνθρωπος ο οποίος είμαι υπεύθυνο για επαφέ με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ποιες είναι οι ουσίες οι οποίες εισάγονται ή φεύγουν από τον κατάλογο των υποψηφίων ουσιών. Κάνουμε δηλαδή ότι ζητούν τα αφεντικά. Αυτή τη στιγμή βέβαια μας είπαν ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, δεν πάβει όμως να είναι πάρα πολύ αργή η πρόοδος. Και αυτό μας ζήτησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών. Ε, είπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Δεν ασχολήθηκα βέβαια τόσο πολύ με τα θέματα ε, προπολογισμού, αλλά να πω ότι η κυρία Χαόπη, η οποία είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα προπολογισμού και κάποιοι άλλοι ε, στην αντιπροσωπεία, εξέφρασαν την έκπληξή τους, ε, διότι φαίνεται ότι ο οργανισμός είναι ικανοποιημένος με αυτό που τους έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϋπολογισμό. Η δική μας εκτίμηση ήταν ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι με τους πόρους που τους διαθέτουν ή που τους έχουν υποσχεθεί ότι θα λάβουν, θα μπορέσουν να διαχειριστούν ε, τον τεράστιο αριθμό καθηκόντων που έχουν, αλλά προς το παρόν δεν ζητούν περισσότερα. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν ε, στο οποίο θα έπρεπε να διαθυπηθεί ε, λίγο περισσότερο η Επιτροπή μας Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα του καταλόγου των υποψηφίων ουσιών και έχω την αίσθηση ότι ίσως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο δραστήριοι ως προς τα θέματα προπολογισμού και πόρων του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έστω και απρόβλεπτη έκθεση. χάρη πιστεύω και στην υποστήριξη από τη φιλανδική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη δουλειά της αυτή η ομάδα του ΕΧΑ, του ΕΚΑ. Έχει καταφέρει ήδη από το πρώτο στάδιο της λειτουργίας του η ομάδα ένα καλό επίπεδο εργασιών και έχει 2,5 εκατομμύρια καταχωρήσει Ηράκλειο έργο έχει επιτύχει να δούμε την επόμενη φάση που πάει με αυτό τον Αύριο το 2010 με 25.000 ουσίες που από ό,τι προβλέπετε θα ε, πρέπει να δηλωθούν, να καταχωρηθούν δηλαδή για πιο προσεκτική παρακολούθηση. Ιδιαίτερος το θέμα του προϋπολογισμού θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί αν δεν έχει υπαρκή πρικοδότηση. Αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει και τη δουλειά της. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το θέμα αυτό υπόψη και τον προπολογισμό του 2011 και να επαγρυπνούμε ώστε να προβλεφθεί η κατάλληλη γραμμή στον προπολογισμό για τη χρηματοδότηση της ΕΚΑ. Και ίσως χρειαστεί να ασχοληθεί και με τα βιοκτώνα. Και η κυρία Κλάς ξέρω ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είναι το επόμενο στάδιο. θεματολογίες με την οποία θα ασχοληθεί η υπηρεσία. Έχουμε συζητήσει αν έχει και το δυναμικό για να το κάνει αυτό και αν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αλλά το λόγο έχει στήσει η κυρία Μαγκίνες παρακαλώ, που ήταν επίσης μέλος προσωπίας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τη συνάδελφο για την ε, προετοίμαστη αυτή έκθεση. Ε, θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η αποστολή για όλους μας. Είδαμε δηλαδή πώς μπορεί ένα νομοθέτημα να αλλάξει την κατάσταση σε ορισμένα θέματα. Ε, θα πρέπει να πω ότι ναι, η Ευρώπη ε, ηγείται των προσπαθειών στον τομέα αυτό, στον τομέα των εργασιών της ΕΧΑ. Έχω κάποιες ενσχέσεις προς τον κατάλογο των ε, συμμετεχόντων. Ίσως έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΚΑ που τελικά δεν είναι δυνατόν να χειριστούμε τα ζητήματα και το πεδίο δραστηριοποίησης όπως θα θέλαμε τουλάχιστον πλευρά της Επιτροπής. Και βεβαίω θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να δούμε τι ρόλο έχουν να διαδραματίσουν όταν υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία χημικών ουσιών ε, καταλόγου ουσιών για παρακολούθηση. Για το φινάλ Α, παραδείγματι, υπήρξε ένα ζήτημα το πλαστικό αυτό για το οποίο υπάρχουν πολλές ε, ανησυχίε. Γιατί, ναι, ακούγονται ε, συχνά ακούει κοινή γνώμη ότι κάποια ουσία μπορεί να είναι επικίνδυνη κτλ. Αλλά μετά ενημερώνεται ότι η υπηρεσία δεν ε, χειρίζεται την ουσία αυτή σαν κατεπήγον σχέδιο. Δεν την εξετάζει δηλαδή με ιδιαίτερη ε, ταχύτητα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, πρέπει να είμαστε θέσει να εξηγήσουμε και στον πολίτη γιατί δεν χορηγείται η προτεραιότητα. Μετά το άλλο ζήτημα είναι βεβαίω οι, ε, που ανταλλάσσουμε, που μοιραζόμαστε με του άλλου κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα και κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, πώ είναι αυτό και επιβλαβέ ακόμη. Αυτό, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ και την ΕΚΑ και του οργανωτέ αυτή τη επίσκεψη που ήταν πολύ χρήσιμη, πιστεύω. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Είχαμε τότε την εντύπωση ότι προχωρεί με πολύ αποφασιστικότητα, ότι είναι στρατευμένη στο έργο της η υπηρεσία αυτή και ότι προσπαθεί να οργανώσει τον συντονισμό αυτό των πληροφοριών, τα ΣΥΦ όπως ονομάζονται. Βεβαίως και υπάρχει ζήτημα όσον αφορά και την διάγνωση των στοιχείων που χορηγούνται, αλλά και τη συνεργασία των κρατών μελών. Επίσης έχουμε προσκαλέσει τον ε, διευθυντή κύριο Ντάντσετ. Ύστερα ίσως από αυτή την ε, πιο καυτή φάση του Νοεμβρίου θα ήταν σκόπιμο να έρθει στην ε, Επιτροπή να δούμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, να μας ενημερώσει για το πώς ε, πάνε αυτές οι εργασίες. Άλλες παρατηρήσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι σας έχω εξαντλήσει όλους με την ψηφοφορία. Καλώς. Θα ξαναλέμε στις 3 ε, πέρας ψηφοφορίας.